Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε σε 7 Ιανουαρίου τον θάνατο του κυρίου Σοάρες, ο οποίος από το 1993 μέχρι το 2004 ήταν ευρωβουλευτής, ανήκε στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ήταν μέλος διαφόρων επιτροπών και πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Στην χώρα του ήταν μια ιστορική προσωπικότητα ο Μάριο Σοάρες. Ήταν σύμβολο της αντίστασης κατά της δικτατορίας και οπωσδήποτε για τους Πορτογάλους και τους Ευρωπαίους συνολικά ήταν ένα σύμβολο για τον αγώνα για την δημοκρατία ως υπουργό Εξωτερικών, Πρωθυπουργό και Πρόεδρος της Πορτογαλίας ήταν μια κεντρική μορφή της δημοκρατικής μεταβολής στην χώρα του και βασικός κινητήριος μοχλός της ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Ευρώπη χάνει έναν μεγάλο πολιτικό άνδρα, έναν οραματιστή και ρεαλιστή, έναν άνθρωπο της αντίστασης στην δικτατορία, έναν μεταρρυθμιστή, έναν αγωνιστή κατά της, του αυταρχισμού και έναν βαθύτατο δημοκράτη. Είναι υποχρέωσή μας να τιμήσουμε την πολιτική του κληρονομιά. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να συλληπιθώ την οικογένεια του Μάριο Σοάρες, ε, τους φίλους του και τους γνωστούς του και σε αυτό το κοινοβούλιο βρίσκονται πάρα πολλοί από αυτούς. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι να σηκωθείτε από τις θέσεις σας προς τη μήνα αυτού του μεγάλου άντρα.